Dear Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Θέλω να σας καλωσορίσω θερμότατα όλους και τους επανεκλεγέντες ευρωβουλευτές από τις διάφορες χώρες, αλλά και τους νέο εκλεγέντες ε, στην Επιτροπή μας με πολύ χαρά χαιρετώ και τα μέλη του προσωπικού, τους διερμηνείς, τους πολιτικούς συμβόλους, όλους εκείνους που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Μιλώ αγγλικά, αν και γερμανίδα, για να ε, με καταλαβαίνετε ε, όσο γίνεται για τα διαδικαστικά. Διότι προεδρεύω εδώ στην πρώτη συνεδρίαση γιατί είμαι απερχόμενη αντιπρόεδρος ε, είναι λίγοι οι εναπομείναντοι συνάδελφοι από την περασμένη θητεία και θα προεδρεύσω μέχρι να εκλεγεί νέος πρόεδρος ή ε, νέα πρόεδρος στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης και θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι θα διαβάσουμε πολλά τώρα για να σεβαστούμε με ευλάβεια την διαδικασία για τη συγκρότηση σε σώμα. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες αυτοί και θα πρέπει να τηρούμε τον κανονισμό όσο γίνεται πιο προσεκτικά. Πρώτον, θα ήθελα να θυμίσω στα μέλη ότι στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι η συγκρότηση ε, του Προεδρίου σε σώμα με εκλογή ενός Προέδρου και ε, τεσσάρων αντιπροέδρων βάσει του άρθρου 204 του κανονισμού. Πρέπει να έχουν οι βουλευτές μαζί τους τις κάρτες ψηφοφορίας, αλλιώς να ζητήσουν τώρα μία ε, κάρτα αντικατάσταση. Δηλαδή, παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε τις κάρτες σας, αλλιώς να σας φέρουμε καινούρια. Ελπίζω να μην χρειαστεί, απλώ να τις έχετε μαζί σας. Αν κάποιος ξέχασε κάρτα, υπάρχει δυνατότητα να ζητήσει αντικατάσταση και μάλιστα πολύ γρήγορα. Μπορούμε να σας βρούμε νέα κάρτα, παρακαλούμε να μας το πείτε. Εάν κάποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του, όχι. Ωραία. Συνεχίζω. Ψηφίζουμε με την εξή σειρά πρώτα τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους. Τα ονόματα των ε, αναπληρωτών που συμμετέχουν είναι ως εξής. Ένας είναι, είναι ο κύριος Ανχέλ Τζαμπάσκι και ζητώ συγγνώμη αν δεν λέω σωστά το όνομά σας. Άγγελ Τζαμπάσκι. Occurs... Σας ε, καλωσορίζω. Αν κάνει κάποια πολιτική ομάδα αλλαγή και ορίσει αναπληρωτή για να ψηφίσει, πρέπει να μας το πει πριν την έναξη της ψηφοφορίας. Δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Ερχόμαστε λοιπόν το κυριότερο σημείο και στην ουσία της συνεδρίασης. Σημειώνω ότι έχουμε απαρτία το 1 τέταρτο των μελών, 7 μέλη. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε και να θεωρηθεί έγκυρη. Τι ε, υποψηφιότητες έχουμε για την εκλογή του Προέδρου. Κύριε Σβέφκα, please. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά και αισθάνομαι και με τεράστια τιμή γιατί ε, θα ήθελα να καλωσορίσω εκ, εκ μέρους του μεγαλύτερου κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ΕΛΚΑ, του νέου συναδέλφους και τις νέες συναδέλφισες. Και θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνεργασία κατά την άρεξη αυτής της κοινοβουλευτική θητείας για την επόμενη πενταετία. Και εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να υποβάλω για τη θέση του Προέδρου της ε, Νομική Επιτροπής για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία τον συνάδελφό μα από την Τσεχία, τον καθηγητή Πάβελ Σφόμποντα. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιβεύκα για την παρουσίαση της υποψηφιότητας και την πρόταση. Ε, σημαντική ερώτηση, κύριε Σφόμωτα. Ε, συνενείτε με την πρόταση αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλος υποψήφιος για τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Uh, Όχι. Ψηφίσουμε λοιπόν. Μπορεί και διαβοής να εκλεγεί ο κύριος Βόμποτα. Αυτή είναι η ταχύτερη και η αποτελεσματικότερη ε, μέθοδος να εκλέξουμε τον νέο μας πρόεδρο. Παρακαλώ όλα τα μέλη που συμφωνούν να γίνει πρόεδρος ο κύριος Σόβοντα να τον χειροκροτήσουμε. Ποιος ζήτησε το λόγο? Ο κύριος Καβαντά, παρακαλώ. Oui, je le cherche. Ήθελα μόνο να σας πω ότι είμαι υπέρ της διαδικασίας εκλογής διαβοής. Uh, that's very nice to hear that you... Καλώς σας. Λοιπόν, Προχωρούμε. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε όσοι θέλουμε να ψηφίσουμε τον κύριο Σφόβοδα για να εκλεγεί πρόεδρος Επιτροπής μας. So, when seen very carefully... Λοιπόν, κοίταξα πολύ προσεκτικά και πρέπει να σας πω ότι κύριε Σφόβοδα έχετε εκλεγεί. Θέλω να σας συγχαρώ εγκάρδια και να σας ευχηθώ να έχετε μια εξαιρετική και επιτυχή θητεία ε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και σας καλώ να έρθετε να πάρετε τη θέση σας και να ε, προεδρεύσετε στην επόμενη φάση. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και είμαι βέβαιος ότι θα περάσουμε συναρπαστικά, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας μου είπαν ότι θα πρέπει να διεκπαιρεώσω γρήγορα το υπόλοιπο της συνεδρίασης και γι' αυτό ακριβώς μιλάω αγγλικά, για να μην χάνουμε χρόνο, περιμένοντας τη διερμηνία. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου μοναδικός αναπληρωτής Α, αποσιάζει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συγκεντρώσει την απαρτία του 1 τετάρτου των μελών, δηλαδή 7 μέλη. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε έγκυρα. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Uh, sorry, I just wanted to tell you the following thing. Uh, Ήθελα να σας πω το εξής. Σε μια συνεδρίαση που είχαμε, σε μια συνεννόηση πριν την έναρξη της συνεδρίασης Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, ε, συμφωνήσαμε οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ να εκλεγώ ως συντονίστρια της ομάδας, της πολιτικής ομάδας, οπότε αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου προτείνω στη θέση μου τη Λίδια Γκέριγκερ. Και Μαντίτελ Βοστέρες, τέταρτον αντιπρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστούμε κυρία Ρέγνερ για την ενημέρωση. Οπότε έχουμε μία υποψήφια για την πρώτη αντιπροεδρία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων την κυρία Λίδια Γκέριγκερ Ντε Ödenberg, αν το λέω σωστά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκέριγκερ, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποψήφια της ε, πολιτικής της ομάδας. Ερωτώ λοιπόν την κυρία Γκέριγκερ, αποδέχεται την υποψηφιότητα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μια και έχουμε μόνο μία υποψήφιο και μία θέση, μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής και πάλι. looking. to up. Yes. Uh, Mrs. Uh, Geringer, would you be so kind and come up and take your seat? Παρακαλώ κυρία Γκέριγκερ, κάντε τον κόπο να έρθετε στη θέση σας στο Προεδρείο. Να περάσουμε τώρα στην εκλογή του δευτέρου αντιπροέδρου. Εξακολουθούμε να έχουμε την απαρτία των 7 βουλευτών, το 1 τέταρτο. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες για τον δεύτερο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Cavada, ε, Um, Περίμενα κάποιον άλλον να προτείνει τη δική μου υποψηφιότητα. Yes, uh, uh, Όπως είχαμε άλλωστε συμφωνήσει και ψηφίσει, αν uh, δεν προθυμοποιείται κανένας, να το προτείνω εγώ. Αλλά ζητώ συγγνώμη να σώσω εγώ από την αμηχανία του συνάδελφου και να τον προτείνω ως υποψήφιο της ομάδας των φιλελευθέρων για τη θέση του Αντιπροέδρου που τη δικαιούται επάξια. Μάλιστα. Άλλος κανείς υποψήφιος? Όχι. Οπότε έχουμε μία και μόνο υποψηφιότητα για τον δεύτερο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ζαν Μαρί Καβαντά. Καταρχήν να ρωτήσω τον κύριο Καβαντά αν συμφωνεί με την υποψηφιότητα. Βέβαια είναι αυτονόητη απάντηση, ρητορική ερώτηση. Αισθάνομαι πολύ πιο άνετα από τη στιγμή που ο συνάδελφος με κατήγγειλε και δημοσίως. Ωραία. Συνενεί ο κύριος Καβαντά. Ας περάσουμε λοιπόν με ψηφοφορία διαβόηση. Thank you very much. Εξελέγει και ο δεύτερος αντιπρόεδρος, τον οποίο και καλό στο Προεδρείο για να καταλάβει τη θέση του. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε για τον τρίτο αντιπρόεδρο της ομάδας, της Επιτροπής Συγγνώμη Νομικών Θεμάτων. Ποιος είναι υποψήφιος? Εκ μέρους του ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά να υποβάλω την υποψηφιότητα του κυρίου Άξελ Βος, πεπειραμένου Ευρωβουλευτή και πολύ καλού φίλου. Μάλιστα, κύριε Βος, Φως, συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σας. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν για τον τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Όχι, περνάμε στην ψηφοφορία διαβοής. Thank you very much and I would like uh, Mr. Foss. Ωραία, κύριε Φως, παρακαλώ, περάστε και εσείς στο Προεδρείο. Και τελευταία εκλογή του τέταρτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες, κυρία Ρέγνερ. Όπως είπα και προηγουμένως, θα ήθελα να προτείνω για τη θέση του τετάρτου Αντιπροέδρου τον συνάδελφο, τη συνάδελφο Μαρή Δελβό Στέρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελβό Στέρες συμφωνεί με την υποψηφιότητά της. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που κατακρεούργησα την προφορά του ονόματός σας. Ωραία. Συμφωνεί η υποψήφια. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για τον τέταρτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Όχι, ας ψηφίσουμε τότε διαβοής. may I ask you also, I would like to ask you to take a seat, but... Παρακαλώ, ελάτε κι εσείς ε, στο Προεδρείο. Yes, please. There is one uh, left for you. Last to announce the next meeting. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Thank you very uh, much for this swift and smooth. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, πολύ εύκολη και γρήγορη ψηφοφορία. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου, 9 το πρωί. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.